περίοδο συνόδου. Τώρα προχωρούμε στην κοινή συζήτηση για την Γεωργία με τη σύσταση του κυρίου Μάμικινς όσον αφορά τη συμφωνία σύνδεσης με την Γεωργία. Κύριε Μάμικινς, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, Έχω την τιμή να ζητάω τη στήριξή σα για την επικύρωση τη Συμφωνία Σύνδεση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γεωργία. Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα. Η Γεωργία και ο λόγο τη Γεωργία πρέπει να αποφεληθούν από νέε ευκαιρίες για να έχουν ένα ευρωπαϊκό μέλλον σταθερό και πετυχημένο. Η Γεωργία ήταν πάντα μια ευρωπαϊκή χώρα. Η κουλτούρα της Γεωργίας αποτελεί μέρος εκείνης της Ευρώπης και σύμφωνα με δημοσκόπηση πάνω από 60% στην Γεωργία στηρίζουν την συμφωνία αυτή. Αυτό σημαίνει βέβαια και μεγάλη ευθύνη από πλευράς των αρχών της Γεωργίας. Η αυριανή επικύρωση είναι συνέχεια του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει αρχίσει εδώ και 8 χρόνια όταν ξεκινήσαμε με το πρόγραμμα δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργίας. Πριν από 5 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες εταίροι άρχισαν με το πρόγραμμα της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Στην αρχή η ολοκλήρωση του έργο αυτού φαινόταν κάτι πάρα πολύ φιλόδοξο. Η Γεωργία όμως φαίνεται ότι πετυχαίνει, κάτι το οποίο δείχνει ότι υπάρχει αποφασιστικότητα από τη χώρα αυτή. Και εξεπλάγει θετικά, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν είδα το έργο που έχει επιτελέσει η κυβέρνηση της Γεωργίας. Δεν ήταν εύκολο να εφαρμοστούν τέτοιες μεταρρυθμίσεις τόσο σημαντικές μέσα σε τόσο μικροχρονικό διάστημα. Είναι δύσκολο να πείσουμε την κοινωνία, τις επιχειρήσεις, τον πολιτικό κόσμο για την αναγκαιότητα γρήγορων μεταρρυθμίσεων. Αλλά ευτυχώς προχωρούν. Οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης μερικές φορές χρειάστηκαν πάνω από 10 χρόνια για να κάνουν τι ίδιε μεταρρυθμίσει, ενώ η Γεωργία μέσα σε λίγα μόνο χρόνια το πέτυχε. Έχει κάνει πολλά μέχρι τώρα. Βέβαια παραμένουν αρκετά ερωτήματα, αρκετά θέματα που πρέπει να προσέξουμε στο μέλλον. Για παράδειγμα, η πόλωση τη κοινωνία, η καταπολέμηση τη διαφθοράς, η Αυχαζία και η Σετία είναι επίσης καυτά ζητήματα. Η Συμφωνία σύνδεση σημαίνει ευθύνη και για τις δύο πλευρές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει τη Γεωργία να καταπολεμήσει την διαφθορά, να έχει ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα, να στηρίξει την ελευθερία του τύπου, να προστατεύσει τις μειονότητες και να κάνει ό,τι μπορεί ο στελός της Γεωργίας να επωφεληθεί πλήρως από την ευρωπαϊκή επιλογή του. Αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να πω εδώ ότι χάρη στη συμφωνία αυτή σύνδεση η Γεωργία περιμένει θετικέ αλλαγέ. Αύξηση εμπορικών συναλλαγών, δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση, διευκόλυνση όσον αφορά το καθεστώ θεωρήσεων, περισσότερε επενδύσει κλπ. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να αποφεληθεί από τη δυνατότητα μεγάλων προγραμμάτων στο εμπόριο, στην ενέργεια, στις μεταφορές και άλλα θέματα στη Γεωργία. Οι επιχειρήσεις δηλαδή ευρωπαϊκές έχουν νέε ευκαιρίες στη Γεωργία. Θα μπορέσουν να επενδύσουν επίσης με ασφάλεια, να αγοράζουν, να πουλούν αγαθά και υπηρεσίες. Εν κατακλείδη, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους που συμμετείχαν στην σύνταξη της έκθεσης αυτής προκειμένου να πετύχουμε την επικύρωση. Θέλω να ευχαριστήσω τους κοιόδους εισηγητές, τους ευρωβουλευτές για τις προτάσεις τους. Ελπίζω, συνάδελφε, ότι η συζήτηση αυτή θα είναι επικοδομητική και θα οδηγήσει σε υιοθέτηση της ε, σύστασής μου. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι Γεωργιανοί αξίζουν θετικές αλλαγές και ελπίζω εμείς οι ευρωβουλευτές να υπερψηφίσουμε τις αλλαγές αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Το λόγο έχει τώρα ο κ. Αβραμόπουλος εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, καταρχάς να ευχαριστήσω εσάς και Αντρέης Βαμίκη για την έκθεσή σας. Μια έκθεση που περιέχει πολλά, πολλές σοβαρές συστάσεις. Δείχνει ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός συνένεσης για την πολιτική μας προς τη Γεωργία. Το Ευρωκοινοβούλιο με την ισχυρή του στήριξη θα μπορούσε να αποστείλει ένα σαφές μήνυμα για την ενίσχυση των δεσμών με την Γεωργία και θα δημιουργούσε εξαιρετικές συνθήκες για στενότερη συνεργασία με τη χώρα αυτή. Η Γεωργία είναι ένας από τους πρωταθλητές στην ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ανατολικής Γειτονίας. Η Συμφωνία Σύνδεσης που κρίνεται αυτή τη στιγμή ε, δείχνει τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και προσδοκίες της Γεωργίας και είναι και το αποτέλεσμα της δικής μας αποφασιστικότητας να χτίσουμε ένα δημοκρατικό σταθερό και ε, δημερό κάτω στην περιοχή με βασική, με βασική σημασία και προτεραιότητα για μας. Η γεωργία θα ε, μεταλλαχθεί εφόσον ε, υλοποιήσουμε την κοινή μα ατζέντα, το κοινό μα θεματολόγιο. Θα προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση εμβαθύνοντα την πολιτική τη σύνδεση και την οικονομική τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γεωργία θα προβλέψει μεταρρυθμίσει που θα επιτρέψουν να ενταχθούν στο δημόσιο βίο ευρωπαϊκέ αξίε, όπω η πολυφωνική δημοκρατία ή ο βαθύτερο σεβασμό των ε, σωστών ε, δικών και του κράτου δικαίου. Η υπογραφή και η προσωρινή ε, θέση σε ισχύ τη συμφωνία θα εξυπηρετήσει και θα διευκολύνει το κοινό Συμβούλιο Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωργία Κάτι που ήδη έγινε ένα μήνα πριν στι Βρυξέλλε προ τη υπογραφή τη συμφωνία, για να δούμε την διαδικασία υλοποίησή τη. Την ίδια ημέρα συμπεράναμε ότι η Γεωργία εκπληρεί τι προποθέσει τη πρώτη φάση αυτού του διαλόγου και σε δεύτερη φάση θα μπορούσε να ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματο δράση αυτό ήταν ακόμα ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία που θα φέρει τη Γεωργία πιο κοντά στο ρόλο της ενός καθεστώτο απελευθέρωση των θεωρήσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, πρέπει να σημειώσουμε ότι η Γεωργία ε, επιτέλεσε σημαντική πρόοδο στις δημοκρατικές της μεταρρυθμίσεις με ανεξάρτητες προεδρικές εκλογές και κοινοβουλευτικές εκλογές το 2012 και 2013 καθώς και εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης το 2014. αλλά και το μήνυμα αυτό ε, απεστάλλει και το ε, αποδέχτηκαν οι Γεωργιανοί, το πολιτικό κλίμα στη χώρα χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση. Οι πολιτικέ αντιπαραθέσει και η πόλωση πρέπει να αποφεύγονται. Πρέπει να βρεθεί χώρο για την αντιπολίτευση και τη διακομματικό διάλογο. Ταυτόχρονα, στο ίδιο πνεύμα, η Γεωργία πρέπει να ε, συνεχίσει τι προσπάθειέ τη για να μεταρρυθμίσει το δικαστικό κλάδο και να βεβαιωθεί ότι επικρατεί κράτο δικαίου στη χώρα. Με μεγάλη χαρά μπορώ να αναφέρω ότι η προσωρινή εφαρμογή της φερικής και σε βάθος συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών από την 1η Δεκεμβρίου ε, ήδη δίνει τα πρώτα της αποτελέσματα. Οι εμπορικές στατιστικές είναι θετικές και σταθερές. Το, ε, ο αντίκτυπος της συμφωνίας βεβαίως αναμένεται ακόμη, όμως οι δείκτες του Σεπτεμβρίου του 2014 δείχνουν 50% αύξηση των εισαγωγών της γεωργίας προς, τους, ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά σε ορυκτά και ε, ξηρούς καρπούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνδράμει τις μεταρρυθμίσεις στη γεωργία και θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας αυτής να προσαρμοστούν στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο με 51 εκατομμύρια ευρώ στήριξη στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος της φετινής χρονιάς, του προγράμματος δράσης. Επιτρέψτε μου τώρα να στραφώ στις προσφατότερες εξελίξεις σε συγκεκριμένε περιοχές της Γεωργίας. Ε, ιδίως την συνθήκη εταιρική ε, στρατηγική σχέση μεταξύ της Ρωσίας και των αρχών της Γεωργίας και του και της Απχαζίας. Βλέπουμε ότι τα πράγματα αλλάζουν, όπως προηγούμενες συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μεταξύ Ρωσικής ε, Ομοσπονδίας και Απχαζίας. Βλέπουμε ότι η λεγόμενη αυτή συνθήκη ε, για την ε, κυριαρχία και την αυτοδιάθεση της Γεωργίας είναι μια αμφισβήτηση. Επίσης, είναι επιζήμια στις διαρκείς προσπάθειες για την σταθεροποίηση της περιοχής και την επικασφάλεια εκεί. Δεν συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης. Επίσης, αντιφάσκει με αρχές του διεθνούς δικαίου και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ρωσική Ομοσπονδία. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, δείχνει αμέριστη στήριξη στην εδαφική κυριότητα της Γεωργίας. Ε, έχουμε δεσμευθεί πλήρως να υποστηρίξουμε την επίλυση διαφορών στη Γεωργία με την συμπροεδρία των, στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και συνομιλίες της Γενέβης και τις αποστολές παρακολούθησης ε, στην Γεωργία επίσης να υπογραμμίσω ξανά την εκτίμηση που πρέπει να εκφράσουμε στη συμβολή της Γεωργίας στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία στα πλαίσια της Συμφωνίας Πλαισίου για τη συμμετοχή της Γεωργίας στις ε, ε, επιχειρήσεις τη κοινή πολιτική άμυνα και ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ολοκληρώνοντα, επιτρέψτε μου να πω ότι η εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Γεωργία είναι ισχυρότατη και θα γίνει ε, αδιάρρηκτη με την ε, έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο της Συμφωνίας Σύνδεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό τώρα ο κύριος Όλι για την Ευρωπαϊκή, ε, από Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου. Πρόεδρε, συνάδελφοι, επίτροπε, η Γεωργία είναι ένας αξιόπιστος εταίρος και έχει επιδιώξει στενότερους πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τις σοβαρές πιέσεις από τη Ρωσία μεταξύ των για ένα μικρό κράτο όπω η Γεωργία, η επιλογή των ελεύθερων συναλλαγών, τη απελευθέρωση του εμπορίου, έχει δώσει καλά αποτελέσματα για τη χώρα την τελευταία δεκαετία. Ε, ο κύκλο εργασιών από τι ε, εξαγωγέ έχει ε, πενταπλασιαστεί ή εξαπλασιαστεί η ανάπτυξη οφείλεται στο φιλελεύθερο καθεστώς ε, της Γεωργίας. Όμως, όπως είπε και ο Επίτροπος, μετά την προσωρινή εφαρμογή της Σφαιρικής και Συμβάθους Συμφωνίας Ελεύθερων Συνολόγων από το Σεπτέμβριο, οι πρώτες ε, στατιστικές δείχνουν τουλάχιστον 50% αύξηση στις εξαγωγές της Γεωργίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, ε, βελτιώθηκε το εμπορικό της ισοζύγιο στη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι, από τους ανατολικούς μας εταίρους η Γεωργία έχει κάνει τις περισσότερες προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση της οικονομίας της και για να ε, εκπληρώσει τις προϋποθέσεις της συμφωνίας και να φτάσει στην κύρωσή της. Η, νέα φάση, η επόμενη φάση της υλοποίησης είναι να στηρίξουμε τη γεωργία προκειμένου να ε, βελτιώσει ακόμη περισσότερο την κατάστασή της. Ευχαριστούμε. Δύο λεπτά. Κύριος Τέτινα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θέλουμε να επικυρώσουμε τη Συμφωνία Σύνθεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ε, Γεωργία μετά την επικύρωση τη Συμφωνίας με τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Το κείμενο που έχετε μπροστά σα είναι καρπός υπομονετική δουλειά από όλες τις πολιτικές ομάδες νομίζω. Έχουμε πολλέ προκλήσει μπροστά μα Να σα θυμίσω ποιε. Πρώτα απ' όλα προσπαθήσαμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Και ας θυμηθούμε πριν από 20 χρόνια όταν προχώρησε σε προσάρτης Απχαζίας η Ρωσία. Μετά θυμηθείτε τον θάνατο 85.000 πολιτών. Θυμηθείτε μετά το 2008 όπου ο Ρωσικός στρατός κατέλαβε την Νότια Σετία. Τι έγινε στην ε, Τσετσενία παραβιάσεις διεθνούς δικαίου συνεχώς από την Ρωσία με τελευταία την προσάρτηση της ε, Κρυμαίας και τα προβλήματα στην Ανατολική Ουκρανία. Όταν λοιπόν συντάξαμε το κείμενο, είπαμε τα πράγματα με το όνομά του. Στην κατοχή την είπαμε κατοχή. Νομίζω ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα ότι δηλαδή ο ρωσικός στρατός θα συνεχίσει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίζονται τα εγκλήματα. Αν αποτύχουμε να θετήσουμε μια ξεκάθαρη θέση, τότε θα είμαστε και εμείς ένοχοι και θα έχουμε και εμείς ευθύνη. Αν η Ευρώπη είχε καταδικάσει την κατάσταση στην Τσετσενία και στην Απχαζία, τότε δεν θα είχαμε φτάσει στην Ουκρανία. Είναι απόδειξη ότι κατάληξε σε νέα συμφωνία η Ρωσία με την Απχασία. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι η προσάρτηση και κάποιων τμήματων της Γεωργίας που θα συμπεριληφθούν στην Ρωσική Ομοσπονδία. Όταν ε, κάναμε τις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίσαμε ότι το καθεστώς της Γεωργίας έχει εκλεγεί δημοκρατικά αλλά είπαμε ότι πρέπει να συνεχίσουν να σέβονται το διεθνέ δίκαιο. Φλέκενστάιν, 1,5 λεπτό από πλευρά Σοσιαλιστική Ομάδα, κυρία Πρόεδρε. Οι Σοσιαλδημοκράτε καλωσορίζουν τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου και φυσικά και τη Συμφωνία Σύνδεση. Και χαιρόμαστε και προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία με τη Γεωργία. Λέμε επίση αφέστατα ότι οι ρωσικέ απόπειρε μέσω των συμβάσεων με τις κατεχόμενες περιοχές να δημιουργήσουν ε, ταραχές και ανασφάλεια θα πρέπει να καταδικαστούν και δεν θα μας σταματήσουν. Και ευχαριστώ το καθεστώς της Γεωργίας για τον πολύ σωστό και ευφυή τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτές τις συγκρούσεις. Η οικονομική συνεργασία θα είναι ωφέλιμη και για τις δύο πλευρές και η πολιτική συνεργασία θα βοηθήσει να μεταρρυθμιστεί και να σταθεροποιηθεί η χώρα ο λαός της Γεωργίας θα παρατηρήσει ότι κράτος δικαίου, καταπολέμηση διαφθοράς, ανεξάρτητη δικαιοσύνη, διαφανής διοίκηση και πολλά άλλα είναι προς όφελός τους. Και είναι καλό λοιπόν ότι ε, θα έχουμε όπως είναι και με την Ουκρανία και με τη Μολδαβία θα έχουμε λοιπόν μια επιτροπή συνεργασίας που θα προωθεί τον διάλογο και με τη Γεωργία και θα μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε ο ένας τον άλλον. Αλλά πρέπει επίσης να σκεφτούμε τι σημαίνει για την Επιτροπή που υπήρχε μέχρι τώρα. Διότι από μία πλευρά θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία και από την άλλη μεριά το Αζερβαϊτζάν και η Αρμενία. Θα είναι δύσκολο αυτό για μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιούρεκ, δύο λεπτά από πλευρά των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συζήτηση που κάνουμε σήμερα και οι αποφάσεις που θα λάβουμε αύριο φαίνεται να έχουν καθυστερήσει τουλάχιστον μια διετία. Ε, το άνοιγμα της ευρωπαϊκής πορείας της Γεωργίας έπρεπε να έχει γίνει το 2008, πριν, αμέσως μετά την ε, επίθεση της Ρωσίας κατά της Γεωργίας. Αυτό θα ήταν μια ειρηνική απάντηση στις επιθετικές τάσεις και ένα σαφές μήνυμα ότι ε, αυτή η χώρα στα ανατολικά της Ευρώπης μπορεί να συνεργαστεί με τη Δύση και να ενισχύσει τις σχέσεις αλληλεγγύης μαζί μας ε, κάτι που να αναχαιτήσει τις προσπάθειες επιθέσεων των αντιπάλων της. Αυτή η θετική μας αντίδραση θα είχαν ε, προλάβει και τα όσα συνέβησαν στην Ουκρανία. Δυστυχώς, ε, βέβαια συνέβη αυτό πολύ αργά, αλλά όπως λέμε στην Πολωνία, καλή αργά παρά ποτέ. Βεβαίως, κάποιος θα πει ότι τα τελευταία χρόνια Φαίνεται να έχουν παραγωνιστεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αλήθεια είναι, αλλά θα πρέπει και να καταλάβουμε, μια και το συζητήσαμε πρόσφατα ακριβώ σε αυτή την αίθουσα και το ακούσαμε και από τον Πάπα Φραγκίσκο, ότι δεν μπορούμε να τους δώσουμε λιγότερα από όσα μας δίνουν εκείνοι. Αυτό το είδος συλλογιστικής για την ανταλλαγή αξιών και αγαθών σε δεύτερη φάση εκφράζει πραγματικά την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και εκεί βασιζόμαστε. Η αντίσταση της Γεωργίας ε, έναντι των ρωσικών πιέσεων και επιθέσεων, η δημιουργία ενός ανεξάρτητου κυρίαρχου κράτους, ήταν μια πολύ σημαντική συμβολή όχι μόνο στην ε, ε, Ευρώπη αλλά και την ασφάλειά μας. Αν η αλληλεγγύη η αλληλεγγύη μας δεν είναι μια λέξη καινή νοήματος, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι καθήκον μας είναι συστηματικά να υποστηρίζουμε την ανεξαρτησία των χωρών που την ανέκτησαν μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό και στο ψήφισμά μας. Ε, Ευχαριστούμε. Ο κύριος Νάρτ έχει τώρα το λόγο για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε είναι μια συμφωνία στρατηγική σημασία. Πολύ βασικό και σημαντικό. Γιατί λέμε διάφορα πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι η Γεωργία είναι Ευρώπη. Δεύτερον, ότι ως Ευρώπη έχει κάθε δικαίωμα να προχωρήσει στις επιθυμίες της, τις απόψεις της και τους εθνικούς της στόχους και την πλήρη σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του άρθρου 49 της συνθήκης μας. Έπειτα, δεν πρόκειται μια δήλωση χωρίς ουσία, πρόκειται για μια δήλωση που αναφέρει συγκεκριμένες υποχρώσεις και για τη Γεωργία και λέει και τι στραβό κάνει η κυβέρνηση της Γεωργίας σήμερα που έχει μια δικαιοσύνη επιλεκτική και που δεν ανταποκρίνεται πάντα στις προδιαγραφές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα κείμενο το οποίο μιλάει για το σεβασμό της ειρήνης, πολύ βασικό και αυτό, που σημαίνει σεβασμό των συνόρων και άρα καταδικάζει οποιαδήποτε πράξη που μπορεί να πλήξει την ειρήνη, την ασφάλεια, δηλαδή οποιαδήποτε ε, κατοχή, οποιαδήποτε παρουσία ε, στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας, για παράδειγμα, στην Οσετία δεν είναι αντίον κανενός. Δεν ε, πρόκειται για αντίφαση με τα νόμιμα δικαιώματα που έχει οποιαδήποτε χώρα κατά μια χώρα που μπορούμε να την πούμε με το όνομά τη, τη Ρωσία, που μπορεί να είναι μια μεγάλη χώρα, αλλά είναι και ένα μεγάλο φίλο τη ε, Ευρώπη. Γιατί και η Ρωσία είναι Ευρώπη. Συνεπώ, πρόκειται για ένα επιπλέον υλικό που φτιάχνει την Ευρώπη και που έχει σαν στόχο την ειρήνη και δεν πηγαίνει εναντίον κανενός. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό τώρα ο κύριος Σόλτς, εκ μέρους της ΓΚΟΕ, της Ευρωπαϊκής Νοτικής Αριστεράς. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η συζήτηση μας σήμερα, ε, ε, παρά το ότι είναι περίπλοκο το θέμα της συμφωνίας, αγνοεί τα βασικά θέματα του μέλλοντος του λαού. Έχουν 35% ανεργία μέσο εισόδημα 350 ευρώ και γι' αυτό πάνω από ένα τρίτο του πληθυσμού έχει μεταναστεύσει ήδη. Με την Συμφωνία Σύνδεσης ε, οι ελπίδες του λαού της Γεωργίας έχουν μία σαφή κατεύθυνση, αλλά κανείς δεν τους εξήγησε πώς θα γίνουν πραγματικότητα οι ελπίδες τους. Πολύ σύντομα, ή καλύτερα η Κομισιόν πρέπει σύντομα να μας πει πώς θέλει να υπάρξει ανάπτυξη της Γεωργίας, πώς θα δημιουργηθούν καλές θέσεις εργασίας που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια δημοκρατική συμβίωση. Και εμείς πρέπει να πούμε τι εννοούμε. Η Γεωργία επέλεξε την οδό της σύνδεσης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει εμείς να σταματήσουμε να καταδικάζουμε και να υπονομεύουμε την ε, ευέλικτη πολιτική της ε, προσπάθειας διακανονισμού των προβλημάτων που έχει με τη Ρωσία. Εάν ε, περάσει η Γεωργία σε κυρώσεις, τότε θα πρέπει εμείς να τους αποζημιώσουμε για τις ζημιές τους. Έληξε ο χρόνος σα, αλλά μπορείτε να δεχτείτε γαλαζιά κάρτα. Από τον κύριο Μαμίκινς. 30 δευτερόλεπτα έχετε. Ε, ευχαριστώ. Η ερώτησή μου είναι, πιστεύετε πραγματικά ότι η προσέγγιση Γεωργίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να επιλύσουν τα οικονομικά προβλήματα της χώρας. Πιστεύετε πραγματικά ότι η απομόνωση της Γεωργίας θα μπορούσε να είναι επιλογή η καλύτερη επιλογή. Κύριε Σόλτ, 30 δευτερόλεπτα. Πιστεύω ότι με την Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών και την Οικονομική ε, Συμφωνία συνδέονται κάποιες ε, προϋποθέσεις και κάποιοι όροι. Και πώς θα μπορέσει η Γεωργία να ενισχύσει την οικονομία της σε σχέση με άλλους εταίρους εμπορικούς, να ανοίξει μια νέα προοπτική. Συνεχίζουμε την, ε, με τους αγόρτες των ομάδων για τους πρασίνους ο κύριος ε, Μέσεριτς για ένα μισή Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω κυρία Μαμίκινς για την ε, ισόρροπη έκθεση που περιλαμβάνει πολύ καλές και χρήσιμες συστάσεις με τις οποίες η Γεωργία, η κυβέρνησή της και οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για τα θέματα αυτά, για το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας, μπορούν να, να ε, ωφεληθούν. Ε, είναι η στιγμή να γιορτάσουμε. Η συμφωνία σύνδεσης, εφόσον είναι σοβαρές, πρέπει να γιορτάζονται. Και θα πρέπει λοιπόν να γιορτάσουμε και προτείνω να γίνει αυτό αύριο. Θα έλεγα όλοι να στηρίξετε τη συμφωνία σύνδεσης και την έκθεση με την ψήφο σας και να γιορτάσουμε στη συνέχεια. Ε, θα Πρέπει επίση κάποια στιγμή να σταματήσουμε για να δώσουμε το χρόνο στου εαυτού μα να συγχαρούν τι Γεωργιανέ Αρχέ που ήδη προόδευσαν, ε, επέφεραν σημαντικότατε αλλαγέ. Πολλά ακόμη μπορούν να γίνουν. έχει πολλέ προτάσει. Οι προτάσει τα επανέλαβε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα τα επαναλάβω κι εγώ. Ωστόσο, εν τέλει, να πω ότι δεν αφισβητώ τα στατιστικά στοιχεία που ανέφερε ο Επίτροπο, απλώ να έχουμε κατά νου ότι οι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών δεν έχουν να κάνουν με αμοιβαία ε, συμφέροντα μόνο, αλλά έχουν να κάνουν και με το κόστο. Να θυμίσω λοιπόν στον Επίτροπο και σε αυτό το σώμα ότι θα παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά το τι συμβαίνει σε περιφερειακό επίπεδο στη γεωργιακή οικονομία και τον ιστό τη χώρα. Κάθε χρόνο θα ενσκέπτουμε στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Κατάληξε Κατάλτη, εξορμός των Πρασίνων. Τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία μου. Μια καλή... Ήταν πολύ καλή η ε, κίνηση αυτή στο τραπέζι των διεθνών διαπραγματεύσεων, αλλά δεν είναι οι συμφωνίες μόνο ε, ένα ποτήρι που πρώτα βλέπουμε γεμάτο. Θα πρέπει να προσέξουμε να μην πέσει μία σταγόνα νερό από ένα γεμάτο ε, ποτήρι. Εάν κανεί δεν προσέξει επίση, ξεχυλίζει το ποτήρι και πέφτει από το τραπέζι, αλλά δεν τρέχει μετά νερό, αίμα τρέχει. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρώπη θα πρέπει να προσέξει τι κάνει σε αυτό το τραπέζι. Νομίζω ότι ρίχνει άφθονο νερό σε αυτό το ποτήρι ε, με, την, ε, με τον κίνδυνο να προκληθούν σοβαρά προβλήματα. Και παρά τα, τις προπόσεις μας. Θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν χώρα αυτή να σέβεται και τα κριτήρια της Κοπενχάγης και αυτό ισχύει και για αυτή τη χώρα και για τους δικούς μας λαούς και για τη Μολδαβία και για την Ουκρανία και για τους φίλους της Γεωργίας. Δεν μας απασχολεί το πότε αλλά το πώς. Γι' αυτό έχουμε τεράστιες αποβολίες, γι' αυτό δεν θα υπερψηφίσουμε αλλά θα απόσχουμε. Ε, η Ρωσία ε, φαίνεται, μάλλον να φαίνεται, ερχόμαστε όλο και κοντά στην κοκκίνη γραμμή στη σχέση με τη Ρωσία. Οι Ρώσοι προφανώς έχουν σοβαρότατες ευθύνε στη χώρα αυτή, αλλά διαρκώς ε, ε, βλέπουμε να προκαλούνται και η περιοχή αυτή γνωρίζει και μια κλιμάκωση της έντασης. Είμαστε σίγουροι για αυτά που κάνουμε. Είδαμε τις ε, δηλώσεις του κυρίου Ολάντ και του Υπουργού, Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Είδαμε ότι οι κινήσεις μας αυτές ουσιαστικά δημιουργούν μεγάλες, μεγάλους κινδύνους το πρόβλημα δεν είναι μόνο να βλέπουμε τι γίνεται στην οικονομία, αλλά να προλάβουμε και να ε, αποτρέψουμε μια ε, ενδεχόμενη σύγκρουση με άλλα μέσα. Τι ψηφίζουμε σήμερα την, για την ευημερία των Γεωργιανών, για τις σχέσεις μας ε, με τους, με τους εταίρους μας από την άλλη όχθη του Ατλαντικού, που αναζητούν εκατομμύρια καταναλωτές για την αγορά τους, ό,τι και αν κοστίσει αυτό ο κύκλος των εργασιών των πολυεθνικών της άμυνας θα αυξανηθεί. Θα αυξηθεί η ρητορική των, ε, του πολέμου πολλές φορές μπορεί να είναι ελκυστική. Αλλά εδώ δεν θέλουμε να προκαλέσουμε τη Ρωσία. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Γιατί μας, ε, ε, δεν μπορεί να μας θυμώνουν οι αρχές μόνο όταν δεν μας βολεύουν. Θα πρέπει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να αναλάβουν εδώ τις ευθύνες τους. Όχι μόνο ο πρόεδρος Ομπάμα από τον οποίο ζητούμε να κρατήσει μια σταθερή στάση. Μετά το Βερολίνο υπήρξαν κάποιε προποθέσει για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Τώρα οι Ηνωμένε Πολιτείε φαίνεται να τα τραβάνε τα άκρα ακόμη, πιο, ακόμη περισσότερο προ τα ανατολικά. Φαίνεται ενδεχομένω εδώ να οδεύουμε προ ένα μοιραίο σφάλμα. Θα έλεγα πάντω ό,τι και αν γίνει να φροντίσουμε να μην χάσουμε, διότι ίσω ήρθε η στιγμή να αλλάξουμε γνώμη και να μεταβάλουμε την πορεία μα. Ευχαριστώ για ένα λεπτό στον ε, κύριο Σόπραντ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, με αυτή τη Συμφωνία Σύνδεσης η Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει ένα νέο κατόφλι σε σχέση με τον ε, περιγυρό τη. Σε δύο σημεία μπορούμε να συνοψίσουμε αυτή τη συμφωνία. Πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται όλο και φτωχότερη. Καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014 δεν είχε ΑΕΠ κατά, α, ε, κατά κεφαλή υψηλότερο από ό,τι στο παρελθόν. Έχουμε μια απώλεια κατά 12% σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για, το, ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών έχει μία μισή φορά μεγαλύτερο ΑΕΠ κατά κεφαλή από ότι ένας Ευρωπαίος. Η σύνδεση με τη Γεωργία και την ε, Μολδαβία θα κάνει ακόμα και πιο φτωχή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, έχουμε όλο και μεγαλύτερα ρήγματα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Είμαστε δίπλα στη Ρωσία, η οποία έχει τα δικά της συμφέροντα, έχει τη δική της σφαίρα συμφερόντων και επιρροής. Η συνεχής επέκταση του ΝΑΤΟ είναι ένα σφάλμα το οποίο θα το πληρώσουμε και το πληρώνουμε ήδη. Οι Ουκρανοί, οι Μολδαβοί και οι Γεωργιανοί δεν πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι θα καθορίσουν το μέλλον της Ευρώπης. Η προσέγγιση της προς το ΝΑΤΟ ή προς τη Ρωσία είναι κάτι το οποίο μπορεί να τους οδηγήσει σε εσωτερικές ε, διαμάχες ακόμα και εμφύλιο πόλεμο. <clears throat> Τα συμφέροντα λοιπόν της Γαλλίας και της Ευρώπης μας οδηγούν να καταψηφίσουμε αυτό το σχέδιο. Ευχαριστώ. Καθίστε όμως έχετε δύο μπλε κάρτες, τις δέχεστε. Η κυρία Καλνιέτε πρώτα. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω τον Γάλλο συνάδελφο το εξή. Μιλήσατε πόσο μας κόστισε η διεύρυνση και πόσο φτωχή είναι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνειδητοποιείτε ότι αυξήθηκε κατά ε, ένα δις η ευρωπαϊκή αγορά. Δηλαδή μπορούν οι επιχειρηματίες σας από τη Γαλλία και από άλλες χώρες να έχουν έξτρα κέρδη. Κύριε Σοπράτ, 30 δεύτερα για να απαντήσετε. Ε, κυρίως συνειδητοποιώ ότι υπάρχει αποβιομηχάνηση και απώλεια για τη γαλλική οικονομία και για πολλές πιο ανεπτυγμένες χώρες. Είναι προφανές ότι όταν ε, ε, εντάσσει στην Ένωση πολλές φτωχές ε, χώρες και είναι πανάκριβη η διαδικασία να ευθυγραμμιστούν, όπως έγινε με τη Γερμανία άλλωστε μετά την επανένωση, ε, τότε αυτό βαρύνει τους πολίτες ε, της πιο πλούσιας Ευρώπης και είναι πάρα πολύ βαρύ το φορτίο και το κόστος. Δεύτερη μπλε κάρτα, ο κύριος Γιούρεκ, 32. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Σοπράτ. Να περιμένω να βάλετε τα ακουστικά σας για να με καταλάβετε. Αγαπητές συνάδελφοι, συνειδητοποιείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερεί και είναι τα ίδια της στα χέρια λόγω της νομισματικής ένωσης. Το κόστος της νομισματικής ένωσης είναι πολύ ψηλότερο από ότι το κόστος της ίδιας της διεύρυνσης. Πραγματικά έχουμε βελτιώσει την οικονομική κατάσταση στην Ένωση με τη διεύρυνση. Απάντηση. Καταρχάς, εγώ θεωρώ ότι η Γεωργία είναι ευρωπαϊκή χώρα από πλευρά ταυτότητα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά πριν τι ελεύθερε συναλλαγέ είχαμε σχέση. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε ανεπτυγμένε συμφωνίε, σύνδεση ελευθέρων συναλλαγών για να έχουμε συναλλαγέ απλέ. Απλώ λέω ότι οι χώρε τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη σήμερα χρειάζονται προστασία στην οικονομία του. Βεβαίω, είναι πολύ ψηλό το νομισματικό κόστο, αλλά και, αυτό εμείς το ε, καταπολεμήσαμε. Συνεχίζουμε. Κύριο Πρέντα, για δύο λεπτά, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ εντυπωσιάζομαι πάντοτε όταν ακούω εδώ και χτες επίσης ακούστηκε η άποψη της Μόσχας που εκφράζεται με μέγα ρητορικό ενθουσιασμό. Μεταξύ άλλων, κύριε Σοπράντ, κάνετε λάθος όσον αφορά τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ για τις χώρες στις οποίες αναφέρετε. Η Μολδαβία δεν θέλει καν να μπει στο ΝΑΤΟ. Κατασκευάζεται μια ιστορία που είναι αυτή που σας διηγούνται οι φίλοι σας, που αν κατάλαβα καλά, διαβάζοντας τον τύπο, σας έδωσαν και χρήματα για το κόμμα σας, έτσι δεν είναι. Το Front National, το είδαμε όλοι στον τύπο, χρηματοδοτείται από τη Μόσχα. Και πραγματικά μα σοκάρει να βλέπουμε και να ακούμε αυτέ τι απόψει. Ξέρω, ξέρω, θα πείτε ότι ε, τα δάνεια είναι δυνατά μέσα στην Ευρώπη. Ε, εντάξει. Αλλά κύριε Σοπράντ μου, ε, στη Γεωργία όπως και στην Κισινάουα στην Μολδαβία και στο Κίεβο στην Ουκρανία οι άνθρωποι έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια ελεύθερη κοινωνία μια κοινωνία ελεύθερων συναλλαγών και την Σοβιετική Αρχή. Από ό,τι φαίνεται αυτού του είδους η Σοβιετική Αρχή σας αρέσει, όπου αποφασίζουν για τους άλλους. Οι λαοί της Γεωργίας, της Μολδαβίας, της Ουκρανίας θέλουν να αποφασίζουν οι ίδιοι και να μην αποφασίζει η Μόσχα για λογαριασμό τους και έχουν το δικαίωμα να ε, ε, σκέφτονται μέσα στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Προοπτική. Τώρα, άμα θέλετε να κάνετε πόλεμο στους καημένου, του Μολδαβού, Γεωργιανού και Ουκρανούς, δεν είναι εδώ το κατάλληλο χώρο. Εδώ είμαστε σε μια λογική αλληλεγγύη και γι' αυτό ακριβώ και η ομάδα του ΕΛΚΑ με ενθουσιασμό θα υπερψηφίσει τη Συμφωνία Σύνδεση όπω το έπραξε για τη Μολδαβία αλλά και για την Ουκρανία. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας ε, μπλε κάρτα τον κύριο Σοπράντ. Τη δέχεστε. No, bien sûr. Βεβαίως, βεβαίως. βεβαίως, χωρίς κανένα πρόβλημα, λέει ο κύριος Πρέντα. Dans cette euh, assemblée, cher Αγαπητέ, ε, κύριε δεν θα πρέπει να παραπληροφορείτε τους συναδέλφους σας. Δεν λάβαμε χρήματα από τη Μόσχα. Ένα δάνειο πήραμε από μια ιδιωτική τράπεζα. Διότι ε, είμαστε απολύτως ελεύθεροι να δανειζόμεθα. Και μέχρι αποδείξη στο αντιθέτου δεν είναι δωρεά το δάνειο. Θα πρέπει να το αποπληρώσουμε σε ιδιωτική τράπεζα, επαναλαμβάνω. Δεύτερο, αγαπητέ κύριε, όταν υπερασπίζεστε μία άποψη ε, αμερικανική σκοπή, δεν σας κατηγορώ ότι είστε πράκτορα τη Ουάσιγκτον. Έχετε το δικαίωμα να έχετε τη γνώμη σας και εγώ τη δική μου. Και μιλούμε εξ ονόματος του ενδιαφέροντος της Γαλλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε κύριε Πρέντε, Επίσης μια, κίτρινη, μια μπλε κάρτα από τον κύριο Καρίμ. Τη δέχεστε. Ορίστε κύριε Καρίμ. Uh, κύριε Πρέντε, θα είμαι υπόχρεος που δεχτήκατε την μπλε κάρτα γιατί θίξατε ένα πολύ. Εδώ υπάρχει ένα σχήμα ε, ρητορική που προέρχεται από ακροδεξιές ε, εξτρεμιστικές ομάδες που πηγαίνουν στα ρωσικά μέσα και μιλάνε κατά του ΝΑΤΟ αλλά και κατά των ίδιων τους των κρατών. Ε, και αυτό τους μετακινεί και τους μετατρέπει σε υπέρμαχους του Πούτιν. Έχουμε χρήματα που πηγαίνουν από τη Ρωσία σε αυτές τις ομάδες. Και δεν είναι μόνο ένας ηγέτης, αλλά περισσότεροι από ένας που πήγαν και κάναν αυτή τη δουλειά. Μήπως θα πρέπει να κάνουμε έρευνα γι' αυτό. Μπορείτε να απαντήσετε και στις δύο μπλε κάρτες, ε, όντας περιεκτικός. Έχετε το λόγο. Όχι, δεν θα απαντήσω στον κύριο Σοπράτ, γιατί είπα από την αρχή να στείλει το ερώτημά του στον Πούτιν ή στους φίλους του στην ε, ιδιωτική αυτή τράπεζα. Αντίθετα να απαντήσω σε αυτά που είπε ο Βρετανός μας συνάδελφος ότι βεβαίως ανησυχούμε που βλέπουμε ότι διάφορες επιχειρήσεις που γίνονται με το Front National γίνονται και στη Μολδαβία. Ένα μολδαβικό κόμμα είχε μπει στην διαδικασία με χρήματα ε, από ιδιωτικέ τράπεζε και ναι, για να κάνει την εκστρατεία του. Είναι απαράδεκτο. Εμεί εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, στο Στρασβούργο και στι Βρυξέλλε, μα δεν είναι εδώ ο χώρο για να εκφράζεται η Μόσχα. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Το λόγο έχει ο κύριο Μποστινάρου για 1,5 λεπτό. Thank Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Ορισμένε φορέ έχουμε την εντύπωση ότι εδώ είναι ορισμένοι σύντροφοι της Μόσχας. Η συμφωνία σύνδεσης με τη Γεωργία δεν είναι ένα βραβείο που δίνουμε, είναι απλώς αναγνώριση της προόδου που έχει επιτευχθεί στη χώρα αυτή, που είναι μια φίλη χώρα. Επίσης, η αναγνώριση της ε, υποστήριξης της κοινή γνώμης της Γεωργίας προς την Ευρώπη. Η κατάσταση βέβαια είναι πολύ, πολύπλοκη στην ε, Μαύρη Θάλασσα και εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο τη γεωργία και σε οικονομικό και σε πολιτικό επίπεδο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τι προσπάθειε αποσταθεροποίηση τη από τη Ρωσία. Όλοι οι φίλοι λοιπόν τη γεωργία θα πρέπει να αγωνιστούν για να υπάρξει μια δικοματική υποστήριξη ώστε να μπορέσει να ευδοκιμήσει η σειρά των μεταρρυθμίσεων που χρειάζονται για να προσεγγίσουν την Ευρώπη νομίζουμε ότι η γεωργία ένα, ένα κομμάτι της, ε, μια ψηφίδα στο παζλ της ε, Μαύρης Θάλασσας όπου η Ρωσία έχει πρόσφατα υπογράψει μια συμφωνία συνεργασίας με την Απχαζία. Αυτό δείχνει την έκταση της παγωμένης σύγκρουσης και φυσικά έχει ακολουθήσει και η κατάληψη αυτής της επαρχίας. Κάτι ακόμα το οποίο θέλω να υπενθυμίσω, τη Συμφωνία Σύνδεσης είναι μια νέα απαρχή. Μια δύσκολη αλλά απαραίτητη εκκίνηση για μια φίλη χώρα, για μια περιοχή που είναι τόσο σημαντική σε στρατηγικό επίπεδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λόγο έχει ο κύριος Τάνοκ για ένα λεπτό. Uh, Κύριε Πρόεδρε, το κόμμα μου, το ECR, λυπάται πάρα πολύ για τη συνεχιζόμενη κατοχή της ε, τμήματος της Ρωσίας από την ε, Ρωσία καταδικάζει την ε, δικαστική δίωξη εναντίον πρώην μελών της κυβέρνησης και του πρώην Προέδρου της Γεωργίας. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η χρονιά αυτή σε ό,τι αφορά τις ε, εταιρικέ σχέσει στο ανατολικό χώρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίω μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Γεωργία. Χαιρετήσουμε αυτή τη συμφωνία γιατί δίνει μια δυνατότητα η Γεωργία να προσεγγίσει πολιτικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίση να ολοκληρωθεί οικονομικά στη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου. Με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας η Γεωργία έχει αναλάβει μια σειρά από υποχρεώσεις να εδραιώσει το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις, σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αστικές ελευθερίες και ενίσχυση των θεσμών της. Πρέπει επίση να ενισχύσουμε περισσότερο τον πολιτικό διάλογο μεταξύ Γεωργία και Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μεγαλύτερη παρουσία τη κοινωνία των πολιτών και μεγαλύτερη ανεκτικότητα έναντι των μειονοτήτων. Είναι λοιπόν γενικά μια καλή συμφωνία που φέρνει τη Γεωργία κοντύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιστέκεται στις πιέσεις της Ρωσίας. Το λέγω έχει ο κύριος Στρεβίσιους για 1,5 λεπτό. Thank you, Mr. President. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι κυρίε και κύριοι, αύριο η έγκριση αυτή της συμφωνίας θα το κάνει μια ιστορική μέρα για την Γεωργία και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχέση των δύο πλευρών. Μια χώρα η οποία είναι στα ανατολικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να τηρεί την ευρωπαϊκή τη προσέγγιση που διαδήλωσε ήδη το 2003. Θέλω να τονίσω την μεγάλη εμπιστοσύνη που έχει δείξει ο λαό τη Γεωργία προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσήλωση τη στην ευρωπαϊκή τη πορεία είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσει <clears throat> να αντιμετωπίσει τι πιέσει που τη ασκεί η Ρωσία η λεγόμενη Συμφωνία Συνεργασίας Ρωσίας-Αφχαζίας είναι ένας τρόπος να δικαιολογήσει το αδικαιολόγητο την προσάρτηση τμήματος του ε, γεωργιανού εδάφους. Δεν δίνουμε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο στην Γεωργία. Έχουμε μπροστά μας ένα Ηράκλειο εγχείρημα το οποίο θα απαιτήσει και από τις γεωργιανές αρχές μεγάλη επιδεξιότητα και ταχύτητα. Το 2015 θα πρέπει να ξεκινήσει η νομική εναρμόνιση με κάπου 1.700 πρωτοβουλίες. Η Γεωργία επίσης θα πρέπει να συνεχίσει τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, να ενισχύσει την οικονομία της αγοράς, να αυξήσει το βιωτικό επίπεδο του λαού της. Εμείς αναμένουμε επίσης από τη Γεωργία να ε, εξασφαλίσει την διαφάνεια και ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδους και να σταματήσει να χρησιμοποιείται εναντίον πολιτικά αντιφρόνοντων. Χρειάζεται μια εθνική συμφιλίωση η Γεωργία και όχι απλώς μια νομική προσέγγιση. νομοθετική προσέγγιση. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ένας εταίρο που θα την υποστηρίξει, αλλά θα είναι και απαιτητικό. Ελπίζω λοιπόν να γίνει πραγματικότητα. έχει για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η Γεωργία καλείται να κάνει μια ελεύθερη επιλογή. Ακόμα και αν ε, το 69% των Γεωργιανών επιθυμούν να υπογραφεί αυτή η συμφωνία και εμείς στο Κοινοβούλιο ε, συμφωνούμε ότι χρειάζεται. Έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος ε, στη δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία της. Απομένει όμως πολλή δουλειά να γίνει δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η προσπάθεια. Δεν θα πρέπει να εμπλέκεται η πολιτική. Είμαι πεπισμένη ότι θα ακολουθήσει το σωστό δρόμο η Γεωργία. Θα πρέπει επίσης να φροντίσουμε να υπάρξει και εμπορική συμφωνία μπορεί οι χώρες να έχουν διαφορετικές λύσεις ή προτάσεις η ε, προτασεις Ορισμένες στρέφονται προς την Ευρασιατική Ένωση και άλλες προς την ε- Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εμπόριο πρέπει να συνεχιστεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Πρόεδρε, θέλω να πω το εξή Στην πολιτική διαδικασία πρόσφατα στη Γεωργία παρουσιάστηκαν προβλήματα στη συνεργασία με την κυβέρνηση. Αυτό μπορεί να είναι ένα καλό ε, παράδειγμα για να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα συζητούμε για την τρίτη ε, συμφωνία σύνδεσης ε, μιας πρώην ε, χώρας κοινοπολιτείας ανεξαρτήτων κρατών. Είναι μια καταπληκτική χώρα η Γεωργία. Έχει κάνει προσπάθειες και έχει πετύχει πολλά στην εσωτερική ασφάλεια. Επίσης έχει δεσμευτεί για την δημοκρατία και την ελευθερία. Για να δούμε εδώ μέσα πώς έχει η δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σηκώνεται ένα συνάδελφο και κατηγορεί άλλου συναδέλφου με πολεμικό τρόπο και επιθετικό που ε, τόλμησαν, άκουσαν, άκουσαν να έχουν διαφορετική άποψη. Ακούστε τι λένε οι πολίτες. Οι πολίτε έχουν κουραστεί και από τη διεύρυνση και από τι συμφωνίε σύνθεσης. Να επανέλθουμε στην αντικειμενικότητα, να σταματήσουμε να επεμβαίνουμε στην περιοχή, να δημιουργούμε ειρήνη και όχι λευκό επιταγέ κάθε μέρα. Ε, είδαμε στην Ουκρανία έχει πέρθει ε, όλεθρος. σχεδόν ε, με τρόπο ιεραποστολικό υπό το μανδύα της αυτοδιάθεσης συνδεόμαστε με τη μία χώρα μετά την άλλη. Οι πολίτες αυτά τα θεωρούν απαράδεκτα. Το λόγο έχει η κυρία Καλνίτε για δύο λεπτά. Mr. President. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αύριο θα επικυρώσουμε τη Συμφωνία Σύνδεσης και θα ήθελα να επαναλάβω το εξής συνήψαμε αυτή τη συμφωνία μετά από έκκληση της Γεωργίας και συμπεριλαμβάνονται εκεί και οι κατεχόμενες περιοχές ε, της Απχαζίας και οι υπόλοιπες. Καλούμε την Ρωσία να τερματίσει την κατοχή αυτών των εδαφών. Είναι μια κοινωνία όπου υποστηρίζει την ένταξη ε, της χώρας κατά πλειοψηφία σε δυτικού θεσμούς και μεταξύ αυτών την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι καθήκον των βασικών πολιτικών θεσμών να εργάζονται συνενετικά στο πνεύμα της Συμφωνίας Σύνδεσης. Θα πρέπει οπωσδήποτε η γεωργιανή κυβέρνηση να μας διαβεβαιώσει και να εξασφαλίσει ότι δεν θα γίνουν επιλεκτικά οι έρευνες και οι διώξεις αντί των πολιτικών τους αντιπάλων. Γνωρίζουμε όλοι ότι η σημερινή αντιπολίτευση είναι ευρενή κυβέρνηση. Αυτό ε, είναι ένα μήνυμα το οποίο επαναλαμβάνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις και αφορά και την πρώην και την ειν κυβέρνηση της Γεωργίας. Το ψήφισμά μας επίσης ορίζει ότι η Γεωργία όπως οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα έχει ευρωπαϊκή προοπτική και μπορούν να υποβάλουν ένταξη αν το επιθυμούν, αίτηση συγγνώμη για ένταξη αν το επιθυμούν. Θα έρθει μια μέρα που η Γεωργία θα είναι τμήμα της διεύρυνσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έχετε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Μάμικινς. Τη δέχεστε. Κυρία Καλνίτε, έχετε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Μάμικινς. Τη δέχεστε. Έχετε μια μπλε κάρτα. You have a blue card from Mr. Mamikins. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Καλνιέτε, εξ όσων κατάλαβα, από το όσα είπατε, εδώ ε, έχετε ε, δύο επιλογές. Είτε η χώρα συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ε, συνεργάζεται με τη Ρωσία. Δεν μπορούμε να φανταστούμε μια κατάσταση όπου μια χώρα μπορεί να είναι μεν ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να έχει και οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία. Um, Απάντησα, κύριε Μαμίκινς. Και βέβαια, η επιλογή μιας χώρας για την ένταξη στην Ευρώπη δεν σημαίνει ότι απομονώνεσαι από τον υπόλοιπο κόσμο. Ας πούμε, δείτε τη Σερβία. Η Σερβία είναι μια χώρα υποψήφια. Έχει λάβει καθεστώς υποψήφιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τη Ρωσία. Βεβαίως είναι μια επιλογή κάθε ε, ξεχωριστής ε, χώρας κυρίαρχη και βέβαια είναι και επιλογή μιας ε, χώρας εταίρου. Ο τρόπος όμως με τον οποίο συμπεριφέρεται η Ρωσία προς τους γείτονές της τους αναγκάζει να επιλέξουν το ένα το άλλο και είναι απαράδεκτο. το λόγο έχει κυρία για λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υποστηρίζω απολύτω την έγκριση της συμφωνίας ε, σύνδεσης με τη Γεωργία. Είναι λογική όσο και απαραίτητη φάση για την ολοκλήρωση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής μεταρρύθμισης από το γεωργιανό λαό. Και το ζητάει ο λαός. Σε ό,τι με αφορά εμένα είναι η αρχή, όχι το τέλος μιας περαιτέρω συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ζητώ ταχεία κύρωση από τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να εμβαθύνουμε την πολιτική συνεργασία και την οικονομική ε, και να γίνει αυτό πραγματικότητα. Είναι σοβαρή η ανησυχία ε, των κρατών μελών και ε, μεγάλες οι προσδοκίες για μεταρρυθμίσεις. Κατοχυρώνεται η ευρωπαϊκή πορεία της Γεωργίας ε, με πολυφωνία στην πολιτική, υπεύθυνη διοίκηση, ανεξάρτητη δικαιοσύνη και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η κυβέρνηση ε, θα πρέπει να είναι προσιλωμένη προς αρχές αυτές ε, και να σταματήσει την πόλωση. Ο μεσαίος χώρος στην κοινωνία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ε, για να επαγρυπνεί, για να γίνουν απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Τέλος, θέλω να σας εκφράσω την ανησυχία μου για την πρόσφατη συμφωνία ε, ολοκλήρωσης Ρωσίας-Απχασίας. Μπορεί να έπεται και η Οσετία. Ε, στις ε, περιοχές η Ρωσία όλο και περισσότερο προελάβνει. Μα να ανησυχεί αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μπέλντερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρον ζήτημα και ερώτημα για το 2015 θα είναι η έκβαση των διεθνών διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αλλά κύριε Πρόεδρε, τι σχέση έχει αυτό με τη σημερινή συζήτηση ε, για τη Γεωργία. Ε, θέλω να είμαι σύντομος. Οι δραστηριότητες εκατοντάδων Ιρανικών επιχειρήσεων στη Γεωργία ε, είναι παράνομες ε, και ε, παρακάμπτουν τις κυρώσεις απέναντι στην Τεχεράνη και ε, θέλουν να ενισχύσουν το πυρηνικό πρόγραμμα. Ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιγόντως ποια βήματα θα κάνετε σε στενή συνεργασία με τις αρχές της Γεωργίας προς τη συνεχιζόμενη προσπάθεια του Ιράν να αυξήσει τα πυρηνικά. Πώς θα ασκήσετε πίεση στο Ιράν στην τελευταία και κρίσιμη φάση διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Λούνατσεκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, όπως είπαν οι συναδελφοί μου, οι πράσινοι υποστηρίζουν αυτή τη συμφωνία <clears throat> εταιρική σχέση και σύνδεση, γιατί υποστηρίζεται και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση και από ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Με αυτή λοιπόν τη συνένεση υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε την πόλωση που υπήρξε στο πολιτικό στερέωμα και να δημιουργήσουμε τις απαραίτητε συνθήκε συμφωνίας μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευσης με ένα τέτοιο τρόπο που θα ξεπεράσει την παραδοσιακή πολιτική αντιπαράθεση. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τις εκρήξεις Ισλαμοφοβίας και ομοφοβίας που έχουν λάβει η χώρα στην Γεωργία και την αδυναμία της δικαιοσύνης να αντιμετωπίσει τους δράστες αυτών των αδικημάτων. Θέλω να θέσω και ένα ερώτημα προς την Κομισιόν. Θα <clears throat> ασκήσετε πίεση στις αρχές της Γεωργίας για τα επενδυτικά σχέδια για σταθμούς ενέργειας και να εξασφαλίσετε ότι θα τηρήσουν τους κανόνες που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος για τέτοιους φορείς. για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ υποστηρίζω την πολύ εντατική εργασία του συναδέλφου για την αυριανή συμφωνία σύνδεσης με την Γεωργία. Ε, έγιναν πολλές ε, συζητήσεις στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Αύριο θα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τη Γεωργία, η αρχή μιας νέας φάσης στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και επικύρωση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας αυτής που είναι μέλος της ανατολικής μας εταιρικής ε, σχέσης, δύο χώρες ε, και ακόμα έχουν ε, ακολουθήσει το παράδειγμα της Ουκρανίας, η Μολδαβία αλλά και η Γεωργία. Δυστυχώς οι χώρες αυτές ε, βρίσκονται σε ένα πλαίσιο παγωμένης σύραξης στην άμεση γειτονία τους, μια σύραξη στην οποία καθηγεί η Ρωσία που προσπαθεί να επιβάλλει τη θέση της και να επιβάλλει στις χώρες αυτές τις επιλογές τους. Στο, το πλαίσιο της σύνθεσης ε, θα ενισχύσει όχι μόνο τις πολιτικές και οικονομικές μας σχέσεις, αλλά θα βοηθήσει και όσον αφορά την κατάσταση της ασφάλειας αυτών των χωρών. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέσο για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το κράτος δικαίου, τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος, αλλά επίσης και πάνω απ' όλα την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος των χωρών. Ε, ως προς αυτό θα ήθελα να συμβουλέψω τους γεωργιανούς συνάδελφους να χρησιμοποιήσουν ε, ειδικού συμβούλους που θα έρχονται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μπορούσαν να τους προσφέρουν την εμπειρογνωμοσύνη τους, γιατί δεν είναι καλό να... Ε, θεωρούμε πως ε, δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται τώρα στη Γεωργία, δηλαδή επιλεκτική χρήση του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης. Ε, ε, ευχόμαστε πολύ θάρρος και καλή επιτυχία στο δρόμο τους. Για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση και είναι ευκαιρία για ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργίας. Η ευρύ αυτή η περιοχή ελευθερου εμπορίου θα έχει ένα σαφές αποτέλεσμα για τους πολίτες της Γεωργίας και τους πολίτες και ένα μεγάλο μέρος των πολιτών υποστηρίζουν την Ευρώπη και αυτό το ποσοστό θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής και στις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει. Ήρθα σε επαφή με τον επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γεωργίας και μαζί του έζησα κάποιες σημαντικές ε, κίνησης προς την εδραίωση της δημοκρατίας και τον κώδικα για τα εργασιακά θέματα και κανόνες για τις επιχειρήσεις και νόμους κατά των διακρίσεων. Αυτή η συμφωνία μου είπε είναι για μας, για τη Γεωργία. Και είναι η ευκαιρία να μπορέσουν να αναγεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ των πολιτικών κομμάτων. Βέβαια παραμένουν σημεία ανησυχία, ιδίω σε ό,τι αφορά για τα θέματα δικαιοσύνη. Πρέπει να μην χρησιμοποιείται το δικαστικό σύστημα ως πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι και η δική μου κυβέρνηση στην ε, Μεγάλη Βρετανία δεν έχει ακόμα συμφωνήσει, ε, δεν έχει ακόμα επικυρώσει την αντίστοιχη η Κροατία είναι η δέκατη χώρα η οποία έχει κυρώσει αυτή τη συμφωνία, αλλά η δική μου χώρα δεν το έχει πράξει. Ελπίζω ότι αυτό θα αλλάξει πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Καρίμ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ω Πρόεδρο τη Αντιπροσωπεία για τον Νότιο Κάφκασο, ε, χαίρομαι που βλέπω πω ο συγητή έχει σπίσει στην ε, ε, παρουσίαση μάλλον στην έκθεση μια σαφή, ε, ένα σαφή προσανατολισμό για το ευρωπαϊκό μέλλον της Γεωργίας. Θα πρέπει να ξέρει η Γεωργία, να γνωρίζει την αλληλεγγύη μας. Η γεωργιανή κυβέρνηση έχει σαφώς έναν σταθερό δρόμο μπροστά τη. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να εφαρμοστούν οι διάφορες μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται από τη Συμφωνία Σύνδεσης. Αναγνωρίζουμε τις πολιτικές προκλήσεις που αποτελούν αυτές οι αλλαγές, αλλά πρέπει να γίνουν η παρακολούθηση της εφαρμογής της Συμφωνίας Σύνδεσης και η βαθιά και καθολική ε, εμπορική συμφωνία ε, ελεύθερου εμπορίου θα πρέπει να ελέγχονται. Ο κοινοβουλευτικό έλεγχο όλη αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να παραμένει επικοδομητικό και έτοιμο να προσαρμοστεί σε οποιασδήποτε μελλοντικέ προκλήσει που μπορεί να προκληθούν από την Ρωσική Ομοσπονδία. Ελπίζω πω αύριο θα έχουμε μια αποφασιστική και ξεκάθαρη ψηφοφορία που θα ε, δείξει την σαφήνεια της θέσης του Ευρωκοινοβουλίου απέναντι στη Γεωργία. Τον κύριο Κάρβερ, τη δέχεστε. Κύριε Κάρβερ, έχετε το λόγο για 30 δεύτερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εσείς ε, ε, έχετε όραμα να επεκταθεί από τον Ατλαντικό στα Ουράλια και πιο πέρα. Τώρα φτάσατε στην Γεωργία, στην Ουκρανία. Πόσο ακόμα θέλετε να πιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που βασίζεται στις αξίες μας είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα εξυπηρετεί όχι μόνο το, τους λαούς της Ευρώπης, αλλά ολόκληρο τον κόσμο. Και ε, το γεγονός ότι εμείς, η χώρα μου και η κυβέρνησή μου, έχουμε ένα όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ισχυρή και ενωμένη και συναποτελείται από χώρε που μοιράζονται κοινέ αξίες, είναι μια εικόνα στην οποία στηρίζει ολόκληρο αυτό το Ευρωκοινοβούλιο και εγώ εγκρίνω και τη θέση του Πρωθυπουργού μου. για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Βουλή της Γεωργίας έχει λάβει θέση σχετικά με ένα νομοσχέδιο για την βελτίωση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γεωργία έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες και αποτελεί σημαντικό βήμα η έγκριση αυτής της συμφωνίας στο δρόμο της προς την ελευθερία. Έχει επιλέξει τον ευρωπαϊκό δρόμο, την ευρωπαϊκή πορεία, γεωργία, παρά τις πιέσεις και τις απειλές που ασκεί η Ρωσία εκεί. Η Ρωσία ε, καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτή η συμφωνία και η Ουκρανία επίσης. Ο πρόεδρος Ποροσέγκο θεωρεί τη Συμφωνία Σύνδεσης με τη χώρα της τη σημαντικότερη φάση της ιστορίας της Ουκρανίας μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Η Συμφωνία Σύνδεσης είναι αποφασιστική σημασία για το μέλλον και πρόκειται για ένα σημαντικό σταυροδρόμι αυτή τη στιγμή. Ποιο δρόμο θα επιλέξει η Γεωργία. Θα στραφεί προς την Ευρώπη, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα τη χειραγωγήσει η Μόσχα. Ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε ε, ε, στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Αύριο καλούμαστε να ψηφίσουμε. Ε, θα επιλέξει το δρόμο του Πούτινγκ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ψηφίσαμε τη συμφωνία με την Ουκρανία και πολλοί εκπρόσωποι μεταξύ αυτών και κάποιος από τη χώρα μου ψήφισε υπέρ του Πούτιν. Για να δούμε τι θα γίνει αυτή τη φορά με τη Γεωργία ορισμένες πολιτικές ομάδες θα συνεχίσουν να ψηφίζουν Πούτιν ή θα ψηφίσουν Ευρωπαϊκή Ένωση και το δικαίωμα της Γεωργίας να αποφασίζει. Ευχαριστώ. κύριος Λιμπεράτσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον εισηγητή μας ε, για την εκθεσή του η οποία έχει ιστορικό χαρακτήρα. Είναι η χρονική στιγμή όπου ένας <clears throat> παρατηρητής θα πει τότε ξεκίνησαν όλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από αυτή τη συζήτηση. Για αυτούς που έχουν αμφιβολίες και οι οποίοι δίνουν διαφορετικές ερμηνείες ή διαφορετικές ιδέες σε σχέση με τα θέματα αυτά σας λέω να άλλη μια χώρα έχει θέσει σαν στόχο της την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να δεχτούν τις αξίες μας θέλουν να ακολουθήσουν το νομικό μας σύστημα την τάξη που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη γεωργία είναι η αρχή μιας μεγάλης προσπάθειας ενός μακρού δρόμου και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να κάνει κανείς όλα αυτά που απαιτούνται για να φτάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει όμως να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχει επιλεκτική δικαιοσύνη στο έδαφος της. Δεν υπάρχει δίπλωμα, δεν υπάρχει δική μας επιλογή μεταξύ Πούτιν και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι απόκειται στους Γεωργιανούς. Αυτοί θα πρέπει να συνεργαστούμε με τη Ρωσία και εκεί μπορούμε να του βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Γεια, για ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, κύριε Αβραμόπουλε, η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γεωργίας συμβάλλει στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας αυτής. Όμως η προσέγγιση της Γεωργίας προς την Ευρώπη πρέπει να εδράζεται στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Θα ήθελα λοιπόν από το βήμα αυτό να καλέσω τις αρμόδιες αρχές της Γεωργίας να σεβαστούν πλήρως τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας που επί εκατοντάδες χρόνια ζει και εργάζεται στη γεωργία. στο πλαίσιο αυτό πρέπει οι αρχές της γεωργίας να φροντίσουν πρώτον για την απρόσκοπτη επιστροφή στις αιστείες τους όσων ελλήνων ποντίων το επιθυμούν δεύτερον για την παράδοση σε αυτούς των σπιτιών τους τα οποία έχουν παρανόμως καταληφθεί από τρίτους τρίτον για την προστασία του δικαιώματος ιδιοκτησίας το οποίο έχουν παρανόμως αποστερηθεί αναμένω αποφασιστική δράση από εσάς κύριε Αβραμόπουλε, άλλωστε διατελέσατε υπουργός εξωτερικών και γνωρίζετε το θέμα αυτό. ευχαριστώ. σας ευχαριστώ. το λόγο έχει ο κύριος Κούκαν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, το 2014 θα πρέπει να θεωρείται ως ένα χρόνος χωρίς προηγούμενο στην πορεία και την πρόοδο της Γεωργίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει υλοποιηθεί η συμφωνία και η υπογραφή της ε, παρά την ασταθή κατάσταση στην περιοχή και εξωτερικές πιέσεις της Ρωσίας. Θα πρέπει εμείς να χαιρετήσουμε όμως πάνω απ' όλα την ισχυρή συνένεση που επικρατεί μεταξύ των γεωργιανών πολιτικών κομμάτων αλλά και μεταξύ του λαού, του πληθυσμού της Γεωργίας. Είναι προσιλωμένη προς τον ευρωπαϊκό δρόμο. Κυρίες και κύριοι αυτή τη στιγμή είναι τόσο εδρεωμένη και αποδεδειγμένη η ευρωπαϊκή τους δέσμευση, εμείς έχουμε χρέος να υποστηρίξουμε τη χώρα αυτή στη στρατηγική της ε, προοπτική. Ακόμα περισσότερο τη στιγμή που η βασική εξωτερική πίεση προέρχεται από τη Ρωσία που εξακολουθεί να κατέχει την Απχαζία και την Νότια Οσετία που είναι περιοχές της Γεωργίας. Ο μεγαλύτερος γείτονας της Γεωργίας μπορεί να αντιτίθεται στις προσπάθειες για μεταρρύθμιση στη χώρα και με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Απχαζία εμείς θα πρέπει να καθησυχάσουμε πιστικά τη Γεωργία ότι είμαστε στο πλευρό της. Η Συμφωνία Σύνδεσης είναι το πρώτο σημαντικό βήμα και η απελευθέρωση ε, της όρησης διαβατηρίων ελπίζω να είναι το επόμενο βήμα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα ορθωθούν εμπόδια στο δρόμο της γεωργίας. Βεβαίως και υπάρχει μια διαδικασία βαθιών μεταρρυθμίσεων ακόμα μπροστά της. Θα είναι δύσκολη, μακρά και περίπλοκη η διαδικασία αυτή. Αλλά μπορεί σίγουρα να διευκολυνθεί από την προσήλωση της γεωργίας ε, την ευρωπαϊκή πορεία. Βεβαίως με τη δική μας ενεργή υποστήριξη και συμμετοχή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Κριστέα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αύριο το Κοινοβούλιο αποφασίζει για την, κύρωση τη τρίτη γενεά τη συμφωνία σύνδεση μετά από αυτήν με την Ουκρανία και τη Δημοκρατία τη ε, Μολδαβία, τη Συμφωνία για την Γεωργία. Η κύρωση αυτή όχι μόνο θα αναγνωρίσει την πρόοδο που έχει γίνει, αλλά και την ε, φιλοδοξία και δέσμευση τη γεωργία στο ευρωπαϊκό μονοπάτι. Η συνυπογραφή συμφωνιών ανάμεσα στην Γεωργία, την Μολδαβία και την Ουκρανία έγινε στι Βρυξέλλε στην ίδια ημερομηνία. Η αυριανή η απόφαση για τη Συμφωνία Σύνδεση με το Γεωργιά ακολουθεί την κύρωση που νωρίτερα ψήφισε φέτο το Κοινοβούλιο μα για την Μολδαβία και την Ουκρανία. Και ολοκληρώνει μια διαδικασία σε αυτό το σώμα, ενώ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τι σχέσει, για την επιθυμία αυτών των τριών χωρών να έρθουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τις προσδοκίες των ε, πολιτών τους. Ε, ελπίζω ε, ότι θα έχουμε την ίδια ισχυρή πλειοψηφία που είχαμε στις πρώτες δύο ψηφοφορίες και καλό τα κράτη-μέλη να γρήγορα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κύρωσης. Πιοτρόφσκι για ένα λεπτό. Μικρόφωνο παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η απόφαση της, των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, εκπληρούν τις προσδοκίες του λαού της Γεωργίας. Εμείς έχουμε νομίζω μια συνένεση ότι ο λαός Γεωργία θέλει να στραφεί προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Όλα αυτά έχουν προετοιμαστεί από του Ευρωπαίου ηγέτε το 2008, τον Λεχ Καζίνσκι, τον Μεντελθόντα και τον κύριο Σαρκοζή. Έχουν δώσει δυνατότητα στη Γεωργία να έχει αυτή την προσέγγιση. Χαιρόμαστε λοιπόν που έχουμε υπογράψει τη συμφωνία αυτή σύνδεση με τη Γεωργία και μεγάλη χαρά θα δω να ευδοκιμήσει αυτή η συμφωνία και με άλλε χώρε όπω η Ουκρανία. Ίσως είμαστε όμως πάρα πολύ περιοριστική σε σχέση με τη Γεωργία. Στο σημείο 45 ζητούμε από τη Γεωργία να εφαρμόσει καθ, κανόνες περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά την ενεργειακή της υποδομή. Μα έχουμε μια ιδιαίτερα νεαρή δημοκρατία. Θα πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι. Εγώ έχει ο κύριος Χόκμακ για δύο λεπτά. Ο κύριος Χόκμακ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, πολλοί ομιλητές πριν από μένα έχουν τονίσει την ιστορική σημασία του βήματος στο οποίο προχωρούμε. Δίνουμε ευκαιρίες και δίνουμε και ένα πλαίσιο στο λαό της Γεωργίας που οδηγεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κάνουμε αυτό σε μια χώρα η οποία βρίσκεται κάτω από συνεχείς απειλές της Ρωσίας με κατοχή του ημίσιος του εδάφους της Γεωργίας από τη Ρωσία. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτές τις πιέσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατυπώσουμε σαφώς τη δήλωση αυτή ότι οποιαδήποτε επίθεση κατά της Γεωργίας από τη Ρωσία είναι εξίσου απαράδεκτη όπως αυτή που βλέπουμε από τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Είναι σημαντικό ότι πρόκειται, πρόκειται για μια ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας, η οποία πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τη Γεωργία και την κυβέρνηση της Γεωργίας να διευκολύνει το ελεύθερο εμπόριο, να υπάρξει συνεργασία, να υπάρξουν επενδύσεις σε πολλούς τομείς. Αυτό σημαίνει ότι η γεωργιανή κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις και να κάνει τα απαραίτητα στο εσωτερικό Τι Σημαίνει, σημαίνει ότι δεν είναι αποδεκτό <clears throat> να υπάρξει επιλεκτική δικαιοσύνη και να χρησιμοποιείται αυτή η επιλεκτική δικαιοσύνη από την κυβέρνηση εναντίον της αντιπολίτευση σήμερα συγχρόνως που προσεγγίζει η Γεωργία την Ευρωπαϊκή Ένωση, η γεωργιανή κυβέρνηση θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι και η κοινωνία της Γεωργίας έρχεται πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Θα πρέπει να ενισχυθεί η κοινωνία των πολιτών στην Γεωργία, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και όλες οι ευκαιρίες που μπορούν να προκύψουν από αυτή τη συμφωνία. Είναι μια ιστορική συμφωνία, αλλά είναι και μια πρόκληση για την κυβέρνηση της Γεωργίας να εγκαταλείψει την επιλεκτική ε, δικαιοσύνη και ευκαιρία να πούμε έξω η Ρωσία από τη Γεωργία. για ένα λεπτό. Θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφό Μαμίκινς. Σήμερα χρειάζεται τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γεωργία όχι μόνο για να μπορέσει να παροτρύνει την δημοκρατική ανάπτυξη και την οικονομική επίσης ε, ανάπτυξη, αλλά και για να στείλει ένα μήνυμα στήριξης ε, στο σύνολο της χώρας για την ε, εδαφική της ακαιρεότητα και για να τη στηρίξει απέναντι στις αποσχιστικές τάσεις. Ωστόσο, αυτό το σχέδιο, αυτή η συμφωνία σύνδεσης είναι σημαντική και για τα δύο μέρη. Ε, η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης είναι πολύ σημαντική. Η συμφωνία σύνδεσης με τη Γεωργία είναι εξαιρετικά σημαντική και ε, δυστυχώς μετά από την προσάρτηση της Κρυμαίας η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας ε, ε, μετατρέπεται σε μια περιοχή συγκρούσεων. Είναι πολύ σημαντική για την περιοχή του Καυκάσου και της Μαύρης Θάλασσας δυστυχώς δεν έχουν σωματωθεί στις κύριες επιθυμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Βαλτική και τα Βαλκάνια. Κύριε Πρόεδρε, η συμπερίληψη και άλλων ευρωπαϊκών κρατών στην εσωτερική αγορά της έρευνας είναι πάρα πολύ ε, σημαντική, ιδιαίτερα όταν γίνονται μεταρρυθμίσεις στις χώρες αυτές και έχουμε κράτους δικαίου, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα ή στρατηγική πρόσβαση ε, προς την ε, Μαύρη Θάλασσα για την προμήθεια φυσικού αερίου, πετρελαίου, αγωγούς κλπ. Πώς όμως αυτή τη τόσο φιλόδοξη συμφωνία βλέπουμε διατυπώσεις του τύπου ένταξη Γεωργίας στο ΝΑΤΟ που όχι απλώς αναφέρουν μια χώρα που δεν έχει σχέση τη Ρωσία ε, αλλά ε, μιλούν και για την εμπλοκή της στον Κάφκασο και στο ρόλο που διαδραματίζει μια τέτοια χώρα απέναντι στη Γεωργία. Για ποιο λόγο και πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να απορεί που η Ρωσία θεωρεί τη συμφωνία αυτή απειλή στα πολιτικά και οικονομικά της συμφέροντα. Αφού μόλις προηγουμένως αναφέρθηκε ε, η συμμετοχή της Γεωργίας στην ε, αμυντική πολιτική ε, με ασκήσεις, γυμνάσια και εκπαίδευση των Γεωργιανών. Παρτουσέλο για δύο λεπτά. Μάλιστα. Έχω την εντύπωση από τη συζήτηση προκύπτει ότι κάποιοι φαντάζονταν ότι εμείς φτιάχνουμε τις συμφωνίες για να προκαλέσουμε τη Ρωσία. Ε, έχουμε συνάψει οικονομικές συμφωνίες με την Ουκρανία και την Ουκρανία, μα δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση χωρών, αλλά όχι μόνο ε, ένωση 28 χωρών, αλλά είναι και μια επικράτεια ελεύθερου εμπορίου που διευρύνεται διαρκώς. Γι' αυτό είναι, είναι σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα ανοίγει τη δυνατότητά τη και προσφέρει τέτοιου είδου συμφωνίε σε μια χώρα που είναι δυτική και που έχει προχωρήσει με ευφυή τρόπο προς τον δρόμο της δημοκρατίας. Αρκεί να θυμίσουμε τις εκλογές που έγιναν σε αυτή τη χώρα το 2012 και το 2013, εκλογές ε, οι οποίες ήταν ομαλές, ε, ήταν δυτικού τύπου εντό εισαγωγικών, ε, συνέβαλαν στο να καταστεί πιστή και ικανή να τηρήσει τις συμφωνίες που έχει κυρώσει. Ε, είναι σαφές πως η πορεία που πρέπει να διανύσει η Γεωργία για να γίνει αξιόπιστη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μακρά. Ε, αλλά είναι σημαντικό να, να δώσουμε το χέρι μας ε, στη χώρα αυτή γιατί είναι σημαντικό να διευρυνθεί η αγορά και πιστεύουμε στην εγκυρότητα της συμφωνίας που συνάπτουμε με αυτή τη χώρα και παραλαμβάνω δεν το κάνουμε για να για να προκαλέσουμε ή να περιφρονήσουμε. Όχι, όπως είπαν κάποιοι. Προχωράμε προς αυτό τον δρόμο με την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, όπου συμμετέχουν όλες οι ανατολικές χώρες για να διευρύνουμε ενδεχομένω την Ένωση και να ε, καταστεί η Ένωσή μας Ένωση των Λαών. Κυρία Μούντι, για ένα λεπτό. Thank you, President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κ. Καραμπασλέλη, ο Πρωθυπουργό τη Γεωργία, αναφέρθηκε στι κοινέ μα αξίε. Οι αξίε αυτέ όμω δεν είναι μοναχά το εμπόριο. Εγώ χαιρετίζω τη Συμφωνία Σύνδεση και την συνέχιση των θετικών σχέσεων μεταξύ Γεωργία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η σύνδεση πρέπει να βοηθήσει να βελτιώσει την ποιότητα τη ζωή όλων των ανθρώπων στη Γεωργία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από αυτή τη συνεργασία θα πρέπει να εργαστούμε μαζί με την κυβέρνηση Γεωργία για να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε στο δρόμο τη προσχώρηση προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ενισχύσουμε τη δημοκρατική διαδικασία, την κοινωνία των πολιτών και να κάνουμε τα απαραίτητα για να υπάρξει και κοινωνική πολιτική η οποία δεν περιέχει νόμου που επιφέρουν διακρίσει. Μόνο η κυβέρνηση της Γεωργίας μπορεί να εδραιώσει αυτό το κοινωνικό υπόδειγμα. Εγώ προσβλέπω στη συνεργασία μαζί τους για να δώσουμε την απαραίτητη υποστήριξη ώστε να επιτύχουμε να εδραιώσουμε αυτές τις κοινές αξίες. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Λαντσμπέργκης για δύο λεπτά. Κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Πρόεδρε, Αύριο με την κήρυξη της Συμφωνίας Σύνδεσης με τη Γεωργία η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ε, την ε, τελευταία φάση που ξεκίνησε στο Βίλνιος πέρσι. Σε τρεις χώρες είχαμε υποσχεθεί να τις φέρουμε πιο κοντά μας αν πληρούν τα κριτήρια. Η Γεωργία ήταν η πρώτη και η πιο δραστήρια ε, στο ευρωπαϊκό μονοπάτι και πλήρωσε πολύ βαρύ τίμημα. Σήμερα όμως θα πρέπει να είμαστε περήφανοι που φτάσαμε σε αυτό το σημαντικό ορόσημο. Ωστόσο, απομένουν κάποιες ανισχυτικές εξελίξεις. Εκείνοι που έβαλαν τα θεμέλια για τον ευρωατλαντικό δρόμο υφίστανται πολιτικές διώξεις και είναι επιλεκτική η δικαιοσύνη. Η σημερινή κυβέρνηση θα πρέπει να γνωρίζει ότι λαμβάνεται αυτό υπόψη πάρα πολύ σοβαρά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Γεωργία θα πρέπει να παραμείνει στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων χωρίς διάβρωση των δημοκρατικών ελευθεριών που χρόνια χρειάστηκαν για να επιτευχθούν. Θα πρέπει να είναι ενωμένη ε, στην ευρωατλαντική τους πορεία, στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου. Μόνο έτσι δεν ε, θα εξατμιστεί ως φρούδα υπόσχεση το όνειρό τους. για 1,5 λεπτό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 η Δύση και το δυτικό πρότυπο στη Γεωργία δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Έχει μακρά ιστορία, έχει οικοδομηθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις της χώρας και τώρα συνεχίζεται. Υπάρχουν ήδη μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει και ο κόσμος πιστεύει βαθύτατα πως είναι μια δική τους επιλογή, η ευρωπαϊκή επιλογή. Σήμερα είναι μια ευκαιρία να βρεθεί η νέα ενέργεια που θα χρειάζεται στα επόμενα στάδια για την επίτευξη του στόχου συμμετοχή στην Ένωση. Αυτό ενώνει τον κόσμο και τους πολιτικούς. Η διαδικασία σύνδεσης ε, έχει να κάνει με την προσαρμογή στα ευρωπαϊκά πρότυπα και για την εξασφάλιση της δικαιοσύνης και του ενός σταθερού κράτους δικαίου ως γενική αρχή. Αυτή είναι η βάση για ένα σύγχρονο κράτος, ένα σύγχρονο κράτος το οποίο δεν είναι μόνο αποτελεσματικό στις δημόσιες υπηρεσίες του, αλλά έχει και μια κοινωνία των πολιτών πολύ ισχυρή και ανεπτυγμένη. Πιστεύω πως στον τομέα αυτό και οικονομικά η Γεωργία θα κινηθεί ακόμη γρηγορότερα. Στον δρόμο της προς το Δύση η Γεωργία θα πρέπει να υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να, να, να συμβουλέψουμε τους Γεωργιανούς σωστά ε, και να, και να προσφέρουμε ε, δυνατότητα μετακίνησης άνευ θεωρήσεων ώστε να μπορέσουν να προοδεύσουν γρήγορα και να αισθανθούν την πρόοδο και οι γεωργιανές, όλες οι γεωργιανές οικογένειες. Όμως η επιλογή θα πρέπει να είναι σαφής ε, ε, ώστε να γίνει κατανοητή από όλους τους εταίρους αλλά και από όσους είναι εχθροί όπως η Ρωσία. Αγαπητοί φίλοι από τη Γεωργία, είστε ισχυροί στην ταυτότητά σας και στη σοφία σας, θα τα καταφέρουμε μαζί. Στη διαδικασία του Catch the Eye έχω δεχθεί τρία αιτήματα. Δίνω το λόγο στον κύριο Μπαλτσέτης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαμίκινς. Ε, η Γεωργία είναι η τρίτη χώρα μετά την Ουκρανία και τη Μολδαβία με την οποία συνάπτουμε τέτοιου είδους συμφωνία σύνδεσης. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συμφωνία αυτή όπως υπόθηκε. Υποστηρίζουμε τη δέσμευση της Γεωργίας να ακολουθήσει την ευρωπαϊκή της πορεία. Γνωρίζουμε ότι η χώρα αυτή γνώρισε πολλές δυσκολίες στο παρελθόν λόγω ακριβώς αυτής της απόφασής της. Γι' αυτό ε, χαιρετίζουμε ακόμα περισσότερο την φιλοευρωπαϊκή της επιλογή. Τώρα ε, χρειάζεται να συσφίξουμε τις σχέσεις μας πολιτικές και οικονομικές με τη χώρα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Πετ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. υποστηρίζω ιδιαίτερα την πορεία της ε, <clears throat> Γεωργίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης, η οποία αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Η εφαρμογή βέβαια θα είναι βέβαια ένα μεγάλο εγχείρημα για τη Γεωργία. Ελπίζω ότι μέσα στο 2015 θα μπορέσουμε να δούμε καλύτερα για τις ευρωπαϊκές προοπτικές της Γεωργίας και άλλες χώρες που βρίσκονται σε προχωρημένες συμφωνίες σύνδεσης η επιτυχή εφαρμογή του σχεδίου δράση για τι προξενικέ θεωρίε είναι πάρα πολύ σημαντική. Μπορεί αυτό να είναι ένα από τα σημεία που θα προέλθουν από την διάσκεψη κορυφή τη Ρήγα. Είναι απαραίτητο να υποστηρίξουμε την κυριαρχικότητα και δαφική ακεραιότητα τη Γεωργία και το δικαίωμά τη να παίρνει δικέ τη αποφάσει για την εξωτερική πολιτική τη και τη πολιτική ασφάλεια τη. Η λεγόμενη συμφωνία ε, συνεργασία μεταξύ τη Ρωσία και τη de facto ανεξάρτητη Αφχασία είναι λόγο για μεγάλη ανησυχία. Υπάρχει ο φόβος ότι τέτοιες δραστηριότητες θα οδηγήσουν σε οριστική προσάρτηση στο τμήμα της Γεωργίας στη Ρωσία. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Κοράου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Εγώ ήθελα καταρχήν να εκφράσω κάποιους προβληματισμούς αφού άκουσα ολόκληρη τη συζήτηση ε, από τους συνάδελφους. Ήθελα να αναφέρω κάποιους ε, προβληματισμούς όσον αφορά αυτή τη Συμφωνία ε, Ελεύθερων Συναλλαγών και Σύνδεσης με την Γεωργία. Συχνά μιλάμε για συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Σήμερα η Γεωργία, χτες στη Βολμολδαβία, η Ουκρανία και ακούω τους συναδέλφους να μιλάνε για ιστορικούς δεσμούς, για θεματικές στιγμές. Μάλλον είναι τι σημαντικέ στιγμέ και εμεί είμαστε υπέρ το να γίνονται σεβαστέ οι αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να τι ασπάζονται και άλλε χώρε. Όμω το θέμα είναι, επειδή είμαστε και λίγο δύσπιστοι απέναντι στη Ρωσία, πώ να μην του προκαλέσουμε, όπω έλεγε ο κύριος ε, Μαρτουσέλο. Αυτή είναι η αίσθηση που δίνεται. Ενώ εμεί θέλουμε να παρουσιαστούμε ω μια μεγάλη ενωτική δύναμη που, έχουν, που έχει ενώσει χώρε που ανάμεσά του έχουν κάνει πολέμου για εκατοντάδε χρόνια. Ίσως μπορούσαμε να το καταφέρουμε αυτό και με τη Ρωσία. Στη διάρκεια παρεμβάσεων δέχτηκα άλλα δύο αιτήματα, ένα και τα τελευταία, με τη διαδικασία του Catch Το λόγο έχει ο κύριος Νάγκη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η προσέγγιση της ε, Γεωργίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντική από στρατηγικής πλευράς για την ευρύτερη περιοχή. Είναι ε, θετικό και για μας. Γι' αυτό είμαι υπέρ αυτής της συμφωνίας σύνδεσης. Θα ήθελα να επισήσω την προσοχή σας στο εξής πολύ σημαντικό θέμα που νομίζω ότι δεν ε, το προσέξαμε πάρα πολύ. Η κατάσταση των μειονοτήτων στη Γεωργία είναι πάρα πολύ κρίσιμη για το μέλλον της χώρας. Παρόλο που υπήρξαν κάποια θετικά βήματα και νομικές κινήσεις υπέρ των μειονοτήτων, ε, παραμένει η δυσπιστία και η καχυποψία ε, στις σχέσεις τους με την ε, πλειονότητα του πληθυσμού. Και αυτό μπορεί να έχει να κάνει με την εδαφική ακαιρεότητα και την κυριαρχία της ε, γεωργίας. Νομίζω ότι δεν το προσέχουμε πάρα πολύ. Δεν θα πρέπει να είναι κανείς μάντης για να καταλάβει ποιες απειλές κινδυνεύουν να διαταράξουν την κατάσταση. Ευχαριστώ. Τέλος, ομιλητής με τη διαδικασία του Catch the Eye, ο κύριος Μπενιφέη για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ, όπως και ο κύριος Κοράου, ήθελα να εκφράσω κάποιες προβληματισμούς μου αφού άκουσα αυτή τη συζήτηση που ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Με εντυπωσίασε ότι κάποιος συνάδελφος Ιταλός από το ΕΛΚ, ο κύριος Μαρτουσέλο, ανεφέρθη στο γεγονός ότι όλα όσα κάνουμε εδώ και αυτή η επιλογή τη συμφωνία σύνδεση θα πρέπει να θεωρηθεί ω μια πρόσκληση ή περιφρόνηση απέναντι στη Ρωσία. Εγώ νομίζω πω αυτό ε, είναι κάτι το οποίο έχω ακούσει και σε άλλε παρεμβάσει και νομίζω πω δεν, δεν τοποθετείται καλά έτσι το θέμα. Εμείς ε, τη συμφωνία της σύνδεσης με τη Γεωργία δεν θα πρέπει να την τοποθετούμε σε αυτήν την οπτική, αλλά σε μια οπτική ε, μεγαλύτερη ισχύω και παρουσίας στην περιοχή ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι μονάχα η ΙΠΑ και η Ρωσία έχουν ε, στην περιοχή αυτή της Μαύρης Θάλασσα και του Καυκάσου στη, στη Γεωργία επιρροή σημαντική. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να, να παίξει ρόλο εκεί και αυτή η Συμφωνία Σύνδεσης μέσω της οικονομίας μας επιτρέπει να ασκήσουμε πολιτικό ρόλο. Και τώρα δίνω το λόγο εξ ονόματο της Επιτροπής στον Επίτροπο κ. Αβραμόπουλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Um, let me start by expressing my to the Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ενδιαφέρον του τους και για τις παρεμβάσεις τους. Η συζήτησή μας επιβεβαίωσαν ότι εξακολουθούμε να προχωρούμε σε βήματα που θα εξασφαλίσουν την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς χαιρετήσουμε όλοι την δέσμευση της ε, Γεωργίας να συνεχίσει με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση αυτών των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των πολιτών της Γεωργίας χωρίς καμία διάκριση. <clears throat> θα πρέπει η διαδικασία δίωξης να είναι διαφανής. Δεν θα πρέπει να έχει πολιτικές ιστεροβουλίε. Και θα πρέπει να εξασφαλίσετε η σωστή διαδικασία. Το ιστορικό της εφαρμογής της εφαρμογής Τη συμφωνίας αυτής θα πρέπει να είναι θετικό. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα υποστήριξη προς τη Γεωργία για να φτάσει τον κοινό μας στόχο να οικοδομήσει μια σταθερή, δημοκρατική και ευμαρή χώρα. θα συνεχίσω τώρα στα ελληνικά προς μήνυ του Πρόεδρου μας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η έγκριση αύριο της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργίας ανοίγει την ευρωπαϊκή προοπτική μιας χώρας που από την ιστορία και τον γεωστρατηγικό ρόλο είναι βέβαιο ότι θα διαδραματίσει επίσης ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ειρήνης συνεργασίας και προόδου για τη γεωργία αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. ανοίγει το δρόμο για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία της γεωργίας που θα στηρίζεται στην αρχή του κράτους δικαίου του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες ενός λαού που αφήνει πίσω του τις δύσκολες εποχές και βαδίζει προς ένα πιο αισιόδοξο ευρωπαϊκό μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Το λόγο έχει ο εισηγητής κύριος Μαμίκινς. Ε, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, κύριε Επίτροπε, κύριε Αβραμόπουλε. Η σημερινή συζήτηση είναι άλλη μια επιβεβαίωση για μένα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την πολιτική αλλαγή στην Γεωργία. Η συμφωνία αυτή ανοίγει νέε προοπτικέ, νέε δυνατότητε, δείχνει την αλληλεγγύη μα με τον γεωργιανό λαό και η η βάση, τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η αλληλεγγύη, πολύ προσφυλή σε μας έννοια τους σοσιαλδημοκράτες. Ε, ε, χρειάζεται λοιπόν μια εταιρική σχέση με τη Γεωργία και αυτή θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν στρέφεται ενάντια καμιάς άλλης χώρας. Στόχος μας είναι η συνεργασία προς αμοιβαίο όφελος. Δεν βοηθάει αυτό μόνο τη Γεωργία αλλά και τις γειτονικές χώρες. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συνεισέφεραν στην προσπάθεια αυτή και ε, ελπίζω αύριο να υπερψηφιστεί και να δείξουμε τη σαφή μας υποστήριξη προς τη Γεωργία. Ελπίζω και ο πρόεδρος της Γεωργίας να παραστεί αύριο στην ψηφοφορία και θα δούμε από εκεί και πέρα τη συνέχεια και την εφαρμογή της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαμίκης και εμείς σας ευχαριστούμε για τη δική σας συνεισφορά διότι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό το έγγραφο που εκπονήσατε και που αύριο θα ψηφίσουμε. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το μεσημέρι. Παρουσία, όπως είπατε, του Προέδρου της Δημοκρατίας της Γεωργίας. Τώρα ακολουθεί ε, η διαδικασία της Χαρτούμ και ε, η πρωτοβουλία για το